και να ξεπεράσουμε εμπόδια, Ανησυχούσαμε κάποια στιγμή ότι δεν υπήρχε κάποιο εύκολο αποτέλεσμα, μια εύκολη λύση που να εξυπηρετεί του στόχου των προτάσεων αυτών, αλλά τελικά τα καταφέραμε. Και το αποτέλεσμα που έχουμε ενώπιον μα είναι πολύ θετικό. Έχουμε έναν βασικό στόχο να προστατεύσουμε αποτελεσματικά του καταναλωτέ, ενώ παράλληλα θα πρέπει να άρουμε τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν για την νέα ψηφιακή αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για πρώτη φορά οι Ευρωπαίοι καταναλωτέ και επιχειρήσει θα είναι σε θέση να βασίζονται σε εν γέννη εναρμονισμένου κανόνε, οι οποίοι θα είναι ειδικά σχεδιασμένοι σχεδιασμένη για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Επίσης δίνονται νέοι κανόνες εγγύσεων, σύγχρονοι, μέσω των δύο αυτών νέων κανονισμών που θα καλύπτουν και τις, τα FEE αγαθά. Θα καλύπτουμε κατά αυτόν τον τρόπο όλο και περισσότερα προϊόντα, τα οποία θα κινούνται από τα FEE κινητά και τα λάπτοψ μέχρι τα ε, νέα προϊόντα διαστεδεμένα στο, που είναι διαστεδεμένα στο διαδίκτυο, όλα αυτά τα νέα προϊόντα που έχουμε, οι νέες οικιακές συσκευές. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι ε, Ευρωπαίοι πολίτε με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μπορεί να αγοράζουν αυτά τα εφη προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προβλέπονται απαραίτητε επικαιροποιήσει για το ψηφιακό περιεχόμενο όλων αυτών των προϊόντων, προκειμένου να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά. Τώρα, και για τι επιχειρήσει όμω, οι δύο αυτέ προτάσει αποτελούν πολύ θετικό βήμα όσον αφορά το ζήτημα τη ασφάλεια δικαίου. Η πρόταση για το ψηφιακό περιεχόμενο προτείνει ένα μεγάλο βαθμό εναρμόνιση και αποτρέπει οποιοδήποτε νομικό κατακρεματισμό, ενώ η πρόταση για τι διαδικτυακέ πωλήσει πάλι προβλέπει ευθυγράμμιση των κριτηρίων συμμόρφωση, καθώ επίση και κοινά κριτήρια επανόρθωση παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνετε ότι μειώνεται όλο το διοικητικό άχθο που θα προέκυπταν είχαμε διαφορετικού κανόνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή κοινού κανόνες κανόνων συμβάσεων που να ισχύουν για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα πετύχουμε μέσω των δύο αυτών προτάσεων. Βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι εδώ στα θεωρία. Φαντάζομαι ότι περισσότεροι αγοράζουν πολλά προϊόντα επιγραμμικά. Νομίζω λοιπόν ότι το θέμα αυτό θα τους ενδιαφέρει όλος ιδιαίτερος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην έχουμε δυσάρεστε εκπλήξει όταν αγοράζουμε στο διαδίκτυο, όταν αγοράζουμε από ένα κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση από κάποιο άλλο κράτο μέλο, γιατί τα πάντα, όπω σα είπαμε, τι δύο αυτέ προτάσει θα είναι εναρμονισμένα. Και αναφέρομαι εδώ πέρα στου ε, συμβατικού κανόνε που θα πρέπει να ισχύουν στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Η ε, συμβουλή μου λοιπόν είναι Σα παροτρύνω μάλλον να αγοράζετε ελεύθερα από το διαδίκτυο, να μην ανησυχείτε και να δείξετε εμπιστοσύνη στι δύο αυτέ προτάσει. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ. Εκ μέρου τη Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων το λόγο έχει η κυρία Χάιντι Χάουταλα για ένα λεπτό παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σα ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφου Φω, Γκέπχαρτ και Αριμόν για το έργο τους ό,τι αφορά τι δύο οδηγίε. Όπως θα θυμάστε, η Επιτροπή Γιούρι, δεν κατάφερε να επιλέξει μεταξύ τη ελάχιστη και της μέγιστη ε, ε, εναρμόνιση Παρ' όλα αυτά έχουμε μια διαδικασία εναρμόνισης. Θα πρέπει να εναρμονίσουμε τους κανόνες μας για την προστασία του καταναλωτή. Και ταυτόχρονα έχουμε θεσπίσει ένα νέο στρώμα διατάξεων προστασίας καταναλωτή για το ψηφιακό περιεχόμενο. Και από πολλές απόψεις ήταν επιτυχημένη η προσπάθεια, γιατί αυτές οι δύο οδηγίες ε, περιλαμβάνουν ένα πλέγμα ε, κανόνων που ενισχύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών ε, μια και ανθεί αυτός ο κλάδος της ψηφιακή παροχή υπηρεσιών. Επίση περιορίζεται ο κατακαιρματισμό ε, της ε, νομοθεσίας περί προστασία των καταναλωτών στα κράτη-μέρη και οι δύο οδηγίε προσδιορίζουν και την ενδιάμεση ευθύνη, ώστε ε, να υποβληθούν ένδικα μέσα κατά προηγούμενου κρίκου αλυσίδα των συναλλαγών. Αυτό είναι ένα σημαντικό τρόπο εξασφάλιση τη αλυσίδα προμήθεια. Εκ μέρους τώρα του, του ΕΛΚ, το λόγο η κυρία Εύα Μαϊντέλ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, μερικές φορές εντοπίζουμε τομείς ο οποίος δεν είναι ε, αναγκαία η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν χρειάζεται να επεβαίνει. Ε, δεν ισχύει όμως αυτό γιατί για τον ψηφιακό τομέα θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να αντιμετωπίσουμε τον ανταγωνισμό μεγάλων αγορών όπως της Κίνας. Θα πρέπει εν τη ενώση να δείξουμε την ισχύ μας και να έχουμε ε, σημαντικούς κανόνες προστασίας του καταναλωτή και στον ψηφιακό κόσμο. Να γνωρίζει ο καταναλωτής που μπορεί να κάνει μια καταγγελία ή να επισημάνει ένα πρόβλημα πάνω από 70 εκατομμύρια πολίτες είχαν πρόβλημα με τη συνδρομή τους, αλλά ένα 10% μόνο έλαβαν αποζημίωση. Η πλειοψηφία των πολιτών δεν ήξεραν πού να αποταθούν για να βρουν το δίκαιο τους ως σκαντισηγήτρια του ΕΛΚ στην Επιτροπή Προστασίας του Καταναλωτού προσπάθησα ε, να συμβάλλω στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Τώρα ποια είναι ξεκάθαρα τα πράγματα που ε, θα πρέπει να αποταθεί κάποιος για να ζητήσει αποζημίωση σε περίπτωση που η ψηφιακή υπηρεσία είναι ελαττωματική. Ευχαριστώ τους εισηγητές για την εξαίρετη συνεργασία που είχαμε. Και Επιτέλους έχουμε οδηγία προστασίας του καταναλωτή που δείχνει μια φιλόδοξη Ευρώπη, μια Ευρώπη που διευκολύνει την καθημερινότητα των πολιτών, που κόπτεται για την προστασία τους, ιδιαίτερα στην ψηφιακή εποχή που βρισκόμαστε. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, το λόγο η κυρία Βυρσινή Ροζιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω το εντυπωσιακό έργο των εισηγητών ε, τι δύο αυτές οδηγίες και κυρίως να επενέσω την κυρία Ευελίν Γκέπχαρτ που πραγματικά έδειξε μεγάλη ικανότητα πειθού στο θέμα αυτό. Τα δύο κείμενα αποτελούν πραγματική πρόοδο και για τους Ευρωπαίους πολίτες και για τους ε, εμπόρους και επικαιροποιούμε τους, ε, τις διατάξεις μας και για τα καταναλωτικά θέματα και λαμβάνουμε υπόψη τις νέες υπηρεσίες και δι' τις διαδικτυακές. Χάρη στη συμφωνία αυτή θα έχουμε εύληπτους κανόνες και για τους Ευρωπαίους πολίτες, εξασφαλίζοντας μια ευθυγράμμιση των κανόνων που ισχύουν για τις πωλήσει αγαθών με τους κανόνες που ισχύουν για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου. Επίσης, πολύ θετικό ήταν το γεγονός ότι καλύπτουμε και κάποιο περιεχόμενο περιλαμβάνεται σε απτά αγαθά. Θα ήταν αδιανόητο να προστατεύουμε μόνο για τα υλικά αγαθά τον καταναλωτή, χωρίς να τον προστατεύουμε για λογισμικά που περιλαμβάνονται στα υλικά αυτά αγαθά και που εξασφαλίζουν την εύρυθμη του λειτουργία. Ε, σε ό,τι αφορά το ψηφιακό περιεχόμενο, η σχετική οδηγία είναι πολύ σημαντική για να, γιατί εναρμονίζει τι ευρωπαϊκέ διατάξει έναν τομέα που μερικέ φορέ δεν υπάρχουν καν εθνικέ διατάξει. Χαιρετίζουμε επίση το γεγονό ότι καταλήξαμε σε συμφωνία για να έχουμε ένα ομοιόμορφο ευρωπαϊκό πλαίσιο σε ένα τομέα που ανθεί. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την πραγματικότητα της κατανάλωσης, συμπεριλαμβάνοντας ε, τις συμβάσεις που περιλαμβάνουν χρηματικό αντίτιμο ή ως αντίτιμο, αντίτιμο την παροχή προσωπικών δεδομένων. Γιατί πολλές ε, τέτοιε συναλλαγές έχουμε σε Και συμβάσεις και καλό είναι που περιλαμβάνονται στο κείμενο και λαμβάνονται υπόψη. Θέλουμε μια πραγματικά ενιαία ψηφιακή αγορά που θα προστατεύει τον καταναλωτή. Αυτή είναι η Ευρώπη για την οποία δίνουμε μάχη. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους του ECR, το λόγο έχει ο κύριος Ντάνιελ Ντάλτον. Παρακαλώ. Uh, Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω του τρει συνεισηγητέ για την εργασία τους. Τον έχουμε μια κοινή δέσμη κανόνων για όσου αγοράζουν ψηφιακό περιεχόμενο υπηρεσία στην Ευρώπη. Προφανώς αυτό διευκολύνει τη ζωή των καταναλωτών και των επιχειρηματιών. Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν το πρώτο το οποίο ενέκρινε τέτοια μέτρα, ενώ άλλα κράτη-μέλη δεν είχαν ανάλογου κανόνε. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει μια ευθυγράμμιση εκατομμύρια Ευρωπαίοι καταναλωτέ σε καθημερινό επίπεδο αγοράζουν ψηφιακό περιεχόμενο, κατεβάζουν ψηφιακέ εφαρμογέ, αγοράζουν προϊόντα διαδικτυατά. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε και τι επιχειρήσει ακένε οι οποίε δραστηριοποιούνται όλο και περισσότερο διασυνοριακά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια να πλαισιώσουμε και του πολίτε εκείνε οι οποίοι θέλουν να ανταλλάξουν κάποια προϊόντα τα οποία είναι ελαττωματικά. Καταλαβαίνετε ότι είχαμε το παράδειγμα μια γαλλική εφημερίδα η οποία επιτρέπει την αγορά ψηφιακού περιεχομένου διαδικτυακά, αλλά, αλλά για περίπτωση αποζημίωση ζητά από του πολίτε να υποβάλουν γραπτό στην αίτηση με τον παραδοσιακό τρόπο. Εκ μέρους των φιλελευθέρων, το λόγο έχει η κυρία Ντίτα Χαράνζοβά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Πιστεύω και εγώ ότι μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα των δύο αυτών νομοθετημάτων, καθότι προσπαθούμε να επεκτείνουμε την ευρωπαϊκή εγγύηση και για τα, αγορά, τα αγαθά τα οποία αγοράζουμε διαδικτυακά. Θεωρώ ότι θα πρέπει να επεκταθεί η χρονική περίοδος που προβλέπεται για την αντιστροφή του βάρους απόδειξης για δύο ολόκληρα χρόνια. Η επέκταση όμως τις εγγύησεις από τα έξι μήνες σε ένα χρόνο αποτελεί από μόνο του μια πολύ θετική εξέλιξη. Και αναφέρομαι στην εγγύηση εκείνη η οποία δεν προποθέτει οποιαδήποτε αιτιολόγηση. Προφανώς οι καταναλωτές χρειάζονται ασφαλή προϊόντα. Αν τα προϊόντα δεν λειτουργούν ε, για ένα χρόνο, καταλαβαίνετε ότι δεν θα πρέπει καν να παρέχονται στην αγορά. Πιστεύω λοιπόν ότι το πιο σημαντικό στοιχείο των δύο αυτών προτάσεων είναι ότι μας φέρνουν πιο κοντά σε ένα, μια ενιαία εργαλειοθήκη, ενιαίο σύνολο κανόνων όσον αφορά το ψηφιακό περιεχόμενο στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό και οι πολίτε και οι επιχειρήσει να γνωρίσουν ότι οι κανόνε θα είναι οι ίδιοι και παντού θα ισχύουν με τον ίδιο τρόπο. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να αγοράζουν από οπουδήποτε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ενιαία αγορά. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εκ μέρου του EFDD, ο κύριο Μάρκο Τσούλο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το ηλεκτρονικό εμπόριο προκειμένου να απτυχθεί χρειάζεται την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, οι οποίοι θα πρέπει να αισθάνονται ότι προστατεύονται όταν αγοράζουν online και όταν αγοράζουν με τον παραδοσιακό τρόπο. Και αυτό ισχύει και για τα υλικά αγαθά και για τα ψηφιακά αγαθά και τις υπηρεσίες. Οι προτάσει για τις δύο αυτές οδηγίες όντως βελτιώνουν την κατάσταση για του ε, καταναλωτές και επίση βλέπουμε ότι προστατεύουμε και τις επιχειρήσεις καθότι δεν δημιουργούμε περαιτέρω διοικητικό άκθο, ιδίω για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει το δικαίωμα επανόρθωσης ή ακόμα και καταγγελίας της σύμβασης ή ακόμα και επιστροφής χρηματικού αντιτίμου. Νομίζω ότι ε, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να προβλέπονται συγκεκριμένοι κανόνες όσον αφορά το κόστος αποζημίωσης μείωση ή αποκατάσταση. Καταλαβαίνετε το κόστο αυτό μπορεί να είναι πολύ υψηλό για κάποιε επιχειρήσει. Βλέπουμε πλέον επίση ξεκάθαρα ότι η αγορά ενό ψηφιακού αγαθού ουσιαστικά συνάδει με την αγορά ενό οποιοδήποτε άλλου κλασικού αγαθού. Καταλαβαίνετε ότι η αγορά, για παράδειγμα, ψηφιακή μουσική αντιστοιχεί ουσιαστικά πλέον στην αγορά ενό απλού συντή. Θα ισχύουν και στι δύο περιπτώσει οι ίδιοι κανόνε. Και προβλέπονται εδώ πέρα συγκεκριμένε ρήτρε όσον αφορά την αντικατάσταση ή την αποζημίωση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί βλέπουμε ότι τα μέτρα αυτά θα αρχίσουν να ισχύουν όλο και περισσότερο και για τα μέσα κοινωνική δικτύωση, καθώ επίση και για όλο το περιεχόμενο, το ακουστικό εκείνο το οποίο μπορεί να βρει κανεί σε ψηφιακέ πλατφόρμε. Νομίζω ότι οι αποφάσει αυτέ είναι πολύ σημαντικέ και για του καταναλωτέ και τι επιχειρήσει. Η κυρία Μιλέν Τροστινσκή έχει το λόγο, εκ μέρου ομάδα CNF. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το επιγραμμικό εμπόριο έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις αυτή την ψηφιακή εποχή και έχει γίνει σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων με νέες ευκαιρίες και για τους καταναλωτές. Βέβαια έχει προκαλέσει και μεγάλη τρευλώσεις ανταγωνισμού ε, μέσω των ε, μεγαθυρίων του ίντερνετ, των μεγάλων επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται τη, την έλλειψη κανονιστικής προστασίας του καταναλωτή. Και μάλιστα, ε, χάρη σε αυτό το κείμενο, ε, λαμβάνεται καλύτερη υπόψη η προστασία του καταναλωτή, προσδιορίζοντας το ψηφιακό περιεχόμενο, και εξασφαλίζοντας την συμμόρφωση των συμβάσεων με τις διατάξεις και δίνοντας εχέγγυα για τις online και τις φυσικές αγορές. Έτσι ενθαρρύνουμε τους παραγωγούς και τους καταναλωτές να παράγουν και να καταναλώνουν λιγότερο αλλά καλύτερα. Επίσης, ε, η ισορροπία του γαλλική νομοθεσία για τι ενοχέ πτυχέ μεταξύ καταναλωτή και ε, πολιτική αγοραστή γίνονται σεβαστέ, κάτι που μα χαροποιεί ε, πέραν της ιδεολογικής υποστήριξης ε, ε, της ε, ενιαίας αγοράς που ξεπερνάει το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον που γνωρίζουμε. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Κάρλος Κοέλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθημερινά στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκατομμύρια πολίτε έχουν πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο και ψηφιακέ ε, υπηρεσίε και καταρτίζουν και συμβάσει γι' αυτό. Βέβαια σε κάποια κράτη-μέλη δεν υπάρχουν σαφεί κανόνε για τι αγορέ ε, ψηφιακού περιεχομένου και υπάρχουν πολλέ και ανομοιόμορφε ε, διατάξει για τι συμβάσει on και offline. Με την έδεσμη μέτρων ενισχύουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών και προσβλέπουμε ένα κοινό πλαίσιο δικαιωμάτων για του πολίτε και τι επιχειρήσει, εξασφαλίζοντα προβλεψιμότητα για όλου και κυρίω για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Έτσι, έρουμε τα βασικά εμπόδια που αφορούσαν το ενοχικό δίκαιο και που παρεμπόδιζαν το διασυνοριακό εμπόριο. Η συμπερίληψη και των πωλήσεων με ε, φυσική παρουσία ήταν σημαντικό. Έχουμε ένα ενιαίο πια πλαίσιο κανόνων για τα καταστήματα με υλική αλλά και με εικονική προστασία, εξασφαλίζοντα ενιαία προστασία για του καταναλωτέ και τι επιχειρήσει. Επίση, γίνονται σεβαστά τα κεκτημένα δικαιώματα των κρατών μελών όπω η ε, Πορτογαλία, που ήταν πιο προηγμένα. Αν δεν γίνονταν σεβαστή η νομοθεσία των πιο προηγμένων χωρών για τα θέματα αυτά θα ήταν ε, άδικο και απαράδεκτο. Θα πρέπει να ενισχύσουμε και όχι να αποδυναμώνουμε την προστασία των καταναλωτών. Γιατί η Ευρώπη των πολιτών που προσπίζουμε έχει το καθήκον να προσπίσει και να εγγυηθεί αυτά τα ε, δικαιώματα. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Λούση Άντερσον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό επίτευγμα για τους καταναλωτές, ε, τις επιχειρήσεις και για το δίκαιο των ε, συμβάσεων. Όπως έχει ήδη υποθεί, είναι πάρα πολύ σημαντική αγορά αγαθών που λειτουργούν με λογισμικό, ειδικά για τους καταναλωτές που βασίζονται σε αναβαθμίσεις του λογισμικού αυτού για να συνδέονται στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα το άρθρο 14 προβλέπει ότι οι επισκευέ ή αντικαταστάσεις ελαττωματικών αγαθών πρέπει να γίνονται δωρεάν. Άλλα θετικά στοιχεία το άρθρο 20 που λέει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να ενημερώνουν τους καταναλωτές για τα δικαιώματά τους. Επίσης, θετικό η αυξημένη έμφαση στην αστική ευθύνη των παραγωγών στο άρθρο 17. Ελπίζω αυτά να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Τέλος, τα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν επευξημένη προστασία σε συγκεκριμένους κλάδους, όπως παραδείγματο χάρη το βραχυπρόθεσμο δικαίωμα απόρριψης ελαττωματικών αγαθών και παροτρύνω τα κράτη-μέλη να το κάνουν. Εν ολίγης πρόκειται για μια οδηγία την οποία αξίζει να ψηφίσουμε και με μεγάλη μου χαρά θα το κάνω. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Αντένας Γκουόγκα. Θέλω να συγχαρώ τους συναδέλφους ε, που εργάστηκαν άοκνα για να τα καταφέρουν και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από τη σκοπιά της ψηφιακής ενίας αγοράς. Το ότι όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα αγαθά που θέλουν να αγοράσουν και ότι έχουμε μια εναρμονισμένη προσέγγιση και χαίρομαι ιδιαίτερως για το ότι ακολουθούμε την οδό της εναρμόνισης. Μας έχει οδηγήσει σε μια επιτυχημένη Ευρώπη. Ω και ηγητής ε, στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων εργάστηκα και εγώ σκληρά με τους ε, συναδέλφους ε, και χαίρομαι για το ότι ακολουθήσαμε ακριβώς το θέμα αυτό της εναρμόνισης για την πώληση αγαθών. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω όλους να στηρίξετε και να υπερψηφίσετε αυτή την πρόταση. Σας ευχαριστώ. Κυρία Κρίστελ Σχαλντεμόζ, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα. Έχουμε μια νίκη ε, για τους Ευρωπαίους ε, καταναλωτές οι οποίοι αγοράζουν όλο και περισσότερα πράγματα στο διαδίκτυο και διασυνοριακά και υπάρχει έτσι και καλύτερη επιλογή και καλύτερες τιμές αλλά δυστυχώς είναι και πάρα πολύ δύσκολο να ξέρει κανείς τι δικαιώματα έχει οπότε με την νομοθεσία αυτή διασφαλίζουμε καλύτερη νομοθεσία για τους ε, καταναλωτές και καλύτερη προστασία θα είναι ευκολότερο να αποφύγουν δύσκολες καταστάσεις είναι πάρα πολύ καλό οπωσδήποτε για τους καταναλωτές αλλά ε, επίσης έχουν και δικαίωμα σε επισκευή αντικατάσταση ελαττωματικών ε, προϊόντων ε, και υπάρχει και πληροφόρηση από τους κατασκευαστές. Οπότε μετά από πάρα πολύ ισχυρή δουλειά και το παρευχαριστώ την κυρία Γκέπχαρτα καταλήξαμε σε μια νίκη για τους πολίτες μας και συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Δάριος Ροζάτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα εξετάζουμε δύο νομοθετικές προτάσεις που θα έχουν κέρια σημασία για την ε, δημιουργία και εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας ε, ψηφιακής ευρωπαϊκής αγοράς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συγκητές μας, κυρίως τον κύριο Άξελ Φως και τον κύριο Πασκάλα Ριμών, για την πολύ ποιοτική ε, εργασία τους. Δύο είναι οι βασικοί μας στόχοι με τις οδηγίες αυτές. Εξασφαλίζουμε τα ίδια δικαιώματα στους αγοραστές ε, που αγοράζουν ε, αγαθά ή υπηρεσίες ε, είτε από καταστήματα είτε ψηφιακά, διαδικτυακά. Επίσης, έχουμε εναρμόνιση των κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μία ομοιογενοποίηση, γιατί αυτή τη στιγμή είναι τόσο κατακαιρματισμένη η, αγορά, η η αγορά που δημιουργεί προβλήματα και δημιουργεί και έλλειψη ασφάλειας δικαίου και για τους καταναλωτές αλλά και για τους επιχειρηματίες και χαίρομαι που με τις ε, εκθέσεις μας το αντιμετωπίζουμε αυτό. Επίσης, ε, φροντίζουμε και για τα δικαιώματα των καταναλωτών και χαίρομαι που η οι σχετικέ εκθέσει πέρα στι αρμόδιε επιτροπέ και θα ήθελα να θεωρήσω του συναδέλφου να του εγκρίνουμε και στην Ολομέλεια. Περνάμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye. Δύο ε, συνάδελφοι θα λάβουν το λόγο μόνο. Πρώτη η κυρία Μιχαέλα Σόιντροβα. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, με ιδιαίτερη χαρά θα υπερψηφίσω τι δύο εκθέσεις γιατί βελτιώνουν τα δικαιώματα του καταναλωτή και ταυτόχρονα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τις ε, επιγραμμικές πωλήσει ε, και για την άνθηση της αγοράς ε, παροχής ψηφιακού περιεχομένου που ανθίζει με ραγδαίους ρυθμούς και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα του καταναλωτή και μια ασφάλεια κατά την αγορά ψηφιακών υπηρεσιών. Θα πρέπει επίσης να διευκολύνουμε και το έργο των παρόχων, των επιχειρήσεων, Χαίρομαι λοιπόν που βρήκαμε πολύ ισορροπημένε λύσει για πολλά τεχνικά ζητήματα και καταλήξαμε σε πολιτική συμφωνία για τι δύο αυτέ νομοθετικέ προτάσει, οπότε μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία ε, των δύο εκθέσεων. Από αυτήν την άποψη θα ήθελα να ζητήσω από την ε, Επίτροπο να δραστηριοποιηθεί περισσότερο στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ε, την οδηγία για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές ιδιαίτερα για τα τρόφιμα. Η κυρία Γκραπίνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όντως, αυτές τις δύο οδηγίες περιμέναμε διακαώς εδώ και πολύ καιρό, γιατί θα βοηθήσουν την ανάπτυξη και την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Από στατιστική άποψη, οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι περισσότεροι καταναλωτές λόγω του κατακαιρματισμένου τοπίου της ψηφιακής ε, αγοράς εφαρμόζουν διαφορετικά κριτήρια και δημιουργείται μια έλλειψη ασφάλειας δικαίου. Τώρα επιτυχάνουμε μια εναρμόνιση, κάτι που θα βοηθήσει και τους καταναλωτές ε, να αγοράζουν πιο εύκολα ε, αγαθά διασυνοριακά, αλλά και τους παρόχους υπηρεσιών ή τους πολιτές να τα διαθέτουν διασυνοριακά. Επίσης θα πρέπει να είναι γνωστά τα ένδικα μέσα τα μέσα επανόρθωσης που έχουν οι καταναλωτές στην διάθεσή τους. Θα ήθελα λοιπόν να σας ε, συστήσω να υπερψηφίσετε αυτές τις διεκθέσεις ε, για να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο την ψηφιακή αγορά. Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση. Τώρα έχει και πάλι το λόγο η Επίτροπος. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, Άκουσα το σύνολο της συζήτησης, όλες τις δηλώσεις που κάνανε οι συγητές και συμφωνώ ότι έχουμε μια εξαιρετική ευκαιρία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί αυτή τη στιγμή να εγκρίνει μια συμφωνία η οποία θα λειτουργήσει υπέρ των καταναλωτών και των επιχειρήσεων παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτό ακριβώς χρειάζεται η Ευρώπη, ιδίως στη χρονική αυτή στιγμή όπου βλέπουμε ότι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο συχνά τίθενται να αμφιβόλο. Γι' αυτό το λόγο σε ενθαρρύνω να εγκρίνετε με την ψήφο σα την πολιτική συμφωνία που είχε επιτευχθεί όσον αφορά τη δέσμη για το ψηφιακό περιεχόμενο και τι υπηρεσίε και να στείλετε κι εσεί ένα χειρό μήνυμα ότι μπορούμε πραγματικά να ανταποκριθούμε στι προσδοκίε των Ευρωπαίων καταναλωτών και επιχειρήσεων. Ότι μπορούν πραγματικά να αποφεληθούν και οι δύο πλευρέ από το νέο ψηφιακό περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμβάλλει έτσι ώστε η δέσμευτη μέτρο να μεταφερθεί γρήγορα στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών κατά αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε στι προκλήσει του νέου ψηφιακού περιβάλλοντο. Ευχαριστώ πολύ. Η συγγήτρια Εύελιν Γκέπχαρτ έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θεωρώ ότι Πράγματι, τώρα που θα ψηφίσουμε, θα ενισχύσουμε την καινοτομία και τον ψηφιακό τομέα, γιατί θα δημιουργήσουμε ασφάλεια δικαίου. Ασφάλεια δικαίου για τους καταναλωτές, για τους εμπόρους και για τους κατασκευαστές. Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, δηλαδή, σε έναν τομέα ο οποίος βρίσκεται σε πάρα πολύ ε, μεγάλη συνεχή κινητικότητα. Έχουμε λοιπόν διατηρήσει τα όσα έχουν επιτύχει τα εθνικά νομικά πλαίσια και έχουμε και μια, ένα νέο διεθνές επίπεδο υψηλής ε, προστασίας. Πρόκειται λοιπόν για προστασία του ψηφιακού καταναλωτή, μια καινοτομία έτσι ώστε να επιτύχουμε το καλύτερο για τους ε, καταναλωτές. Και χαίρομαι που το καταφέραμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακολουθεί ο ο κ. Σαξελφός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους τους ομιλητές. Θα ήθελα να απευθύνω και πάλι έκκληση σε όλους ε, τους συναδέλφους εντός σας Το αποτέλεσμα αυτό των δύο αυτών δίδυμων εκθέσεων περί ψηφιακού περιεχομένου και των πωλήσεων μέσω διαδικτύου να το υπερψηφίσουν γιατί έχουμε καταφέρει να κάνουμε ένα καλό βήμα και στις δύο εκθέσεις ε, και έχουμε επεκτείνει την εγγύηση στα δύο έτη, προχωρήσαμε σε πλήρη εναρμόνιση ε, και αντιστροφή του βάρους αποδείξεως σε ένα διάστημα μεταξύ ενός και δύο ετών. Είναι σημαντικό για την εσωτερική ψηφιακή αγορά και για την νομική ασφάλεια, είναι σημαντικό για τους καταναλωτές και είναι σημαντικό για το διασυναριακό εμπόριο. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν σε αυτό, ιδιαίτερα την ε, Κομισιόν των Πασκάλα και την Εύελιν Γκέπχαρτ βεβαίως για την καλή μας συνεργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και ο, ο Πασκάλα Ριμών επίσης Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, σύντομα πέντε σημεία. Πρώτον, τρία χρόνια σκληρή δουλειά Δεύτερον, πάρα πολλέ συναντήσεις. Τρίτον, πολύ καλή συμβιβασμή. Τέταρτον, ενισχύθηκαν τα δικαιώματα των καναλτών. Πέμπτον, γίνεται ευκολότερη και απλούστερη η ζωή των μικρών επιχειρήσεων. Οπότε ευχαριστώ όλου του συναδέλφου και παρακαλώ να υπερψηφίσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ ολοκληρώνεται η κοινή συζήτηση των δύο εκθέσεων και κερδίσαμε και το τέταρτο που είχαμε μείνει πίσω. Οπότε χωρίς ε, ε, καθυστέρηση μπορούμε να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Ε, σε λίγο θα ψηφίσουμε τις σχετικές εκθέσεις. Μια πολύ σύντομη διακοπή μέχρι τις 12.30.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 Συνεχίζεται η συνεδρίαση. Σας πληροφορώ ότι σύμφωνα με το άρθρο 187 μία ομάδα βουλευτών που μπορεί να φτάσει στο κατώτατο κατόφλι θα υποβάλει αύριο στην αρχή της συζήτησης όσον αφορά τη δέσμη για την κινητικότητα μία ερώτηση η οποία έχει να κάνει με το αποδεκτό, με το αν οι δύο ακόλουθε εκθέσει. Η έκθεση που έχει να κάνει με την πρόταση οδηγία του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 2007 όσον αφορά την εφαρμογή και την συγκεκριμένων μέτρων για την οδηγία 96-2001 καθώς επίσης και την οδηγία που έχει να κάνει με τις οδικές μεταφορές, έκθεση Κίλονεν δηλαδή. Δεύτερον, έκθεση πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό 561 του 2006 όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα που πρέπει να ευσχύουν για την μέγιστη περίοδο οδήγησης σε καθημερινή και εβδομαδιαία επίπεδο, καθώς επίσης και κανονισμός ο οποίος θέτει το κατώτατο επίπεδο ανάπαυσης για τους οδηγούς, καθώς επίσης και την οδηγία εκείνη που έχει να κάνει με την εγκατάσταση ταχυγράφων. Έκθεση Βάντεν Κάμπα. Υπενθυμίζω ότι το θέμα αυτό θα τεθεί αύριο στην αρχή της συζήτησης όσον αφορά τη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα. Πρόκειται για μια ερώτηση που θέτουν ορισμένοι βουλευτές ως προς το αν είναι παραδεκτή οι, παραδεκτές οι δύο αυτές προτάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 187 του κανονισμού μας. Passiamo ora alle votazioni. Ας περάσουμε τώρα στις ψηφοφορίες. Ρέγνερ, όσον αφορά την αίτηση άρσης ασυλίας του Τζον Ντόρμαν. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έκθεση Didier αντιπροσωπευτικέ δράσει για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών. Με νέα ψήφο, μονομαστική κλίση ψηφίσουμε. Άρτη ψηφοφορία, παρακαλώ. Πέρασε. Εγκρίνεται το κείμενο και εγκρίνεται έτσι και η πρώτη ανάγνωση του εκνοβουλίου συγχαρητήρια στον εισηγητή. Περνάμε στην έκθεση Πρέντα, πρωτόκολλο τη Ευρωμεσογειακή Συμφωνία Σύνδεση Ευρωπαϊκή Ένωση Ισραήλ προ χώρε Κροατία. Ψηφίζουμε μονομαστική κλίση, άρτη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρασε. Εγκρίνεται το κείμενο. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Περνάμε στην έκθεση Μακάλιστερ όσον αφορά τη Συνολική Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Ουσμπεκιστάν. Δεν υπάρχει γραπτός καμία ένσταση όσον αφορά τη σύσταση αυτή. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το άρθρο 113, άρθρο 6, εγκρίνεται η σύσταση αυτή. Συγχαρητήρια στον κύριο Μακάλιστερ. Περνάμε τώρα στην έκθεση Ulfstock, τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας. Έχουμε μια πρόταση τροποποίηση τη πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τροπολογή 33 και 34 από κοινού υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχέ. Ηλεκτρονική επαλήθευση, πολύ ωραία. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην πρόταση νομοθετική πράξη. Ψηφίζουμε από κοινού υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνονται. Ψηφίζουμε με μαστική κλίση στο σύνολο τη πρόταση. Άρτη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Το κείμενο εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Περνάμε στην έκθεση Μπούζεκ, Κοινή κανόνε εσωτερική αγορά ηλεκτρική ενέργεια. Ψηφίζουμε την προσωρινή συμφώνια μονομαστική κλίση άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Το κείμενο εγκρίνεται. Δηλώσει επιτροπή. Τροπολογία 201 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Ολοκληρώνεται έτσι πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περνάμε πάλι στην έκθεση και εξωτερική αγορά ηλεκτρική ενέργεια. Ψηφίζουμε την τροπολογία 187, μονομαστική κλίση άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Το κείμενο εγκρίνεται. Περνάμε στη δηλώση επιτροπή. Τροπολογία 188 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ολοκληρώνεται έτσι η πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έκθεση Πέτρεσεν τώρα. Οργανισμό Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Συνεργασία Τροφιμιστικών Αρχών ενέργεια. Προσωρινή συμφωνία. Τροπολογία 91 δηλαδή. Με ονομαστική κλίση άρθρη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρασε. Το κείμενο εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ολοκληρώνεται έτσι και η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Περνάμε στην έκθεση Τζανονάτο. Ετοιμότητα αντιμετώπιση κινδύνων στον τομέα τη ηλεκτρική ενέργεια. Τροπολογία 63 για την προσωρινή συμφωνία. Άρτη ψηφοφορία, παρακαλώ. Ονομαστική κλίση. Πέρας. Το κείμενο εγκρίνεται και ολοκληρώνεται έτσι η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Συγχαρητήρια στον κύριο Τζανονάτο, τον εισηγητή. Περνάμε τώρα στην έκθεση Μπόνη. Σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλε ουσιώδει παραμέτρου. Τροπολογίε Επιτροπή. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνονται. Τροπολογίε τη αρμόδια Επιτροπή 11. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 39. Με ονομαστική κλίση άρτη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 41 σε δύο τμήματα. πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 41. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 53 της Επιτροπής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 62 μονομαστική κλίση άρθρη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21 μονομαστική κλίση άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. πίπτη 63. Περνάμε στροπολογία 22D με ονομαστική κλίση άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. Το κείμενο εγκρίνεται, πίπτη 64, άρθρο 5 σε δύο τμήματα, τροπολογία 58, πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άρθρο 6 παράγραφος 2 τροπολογία 29 D υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται καταπίπτει 65 τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθεια, παρακαλώ Πέρας. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 66, τροπολογία 67, μονομαστική κλίση άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 68 σε τρία τμήματα και τα τρία με το πρώτο τμήμα ονομαστική κλίση. Πέρασε. Απορρίπτεται δεύτερο τμήμα, μονομαστική κλίση. άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται τρίτο τμήμα, άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 μονομαστική κλίση άρτη ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 43. Πολύ ωραία. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 74. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 75. Μονομαστική κλίση. Άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 49. Με ονομαστική κλίση. Άρτη ψηφοφορία. Α, συγγνώμη, έγινε ένα λάθος, λέει ο Πρόεδρος. Υπέρ παρακαλώ, όχι μονομαστική κλίση, ψηφίσουμε κανονικά. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 73, μονομαστική κλίση αυτή τη φορά, άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 59 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Εξήντα με κλίση άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Καταπίπτει 61. Τελική ψηφοφορία για την πρόταση μονομαστική κλίση. Άρτε ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Το κείμενο εγκρίνεται και ολοκληρώνεται έτσι και η πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συγχαρητήρια στον εισηγητή τον κύριο Μπόνι. Παρακαλώ. Επί της ε, διαδικασίας αναφέρομαι στο άρθρο 115 το οποίο αναφέρει ότι θα πρέπει να εργαζόμαστε με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια. Από τις 11 Φεβρουαρίου έχουμε νέες διατάξεις για τη διαφάνεια στους συγητές. Χτες το βράδυ λοιπόν όταν άνοιξα την ε, συνεδρίαση είχαμε συναντήσεις ε, μεταξύ λομπιστών και των εισηγητών της συγκεκριμένης έκθεσης. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω ως πρόεδρος να το διερευνήσετε και να μου πείτε εάν χτες το βράδυ είχαμε συναντήσεις μεταξύ ε, λομπιστών ε, χωρίς παρουσία δημοσιογράφων συγκεκριμένα. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω ε, εξυβρίστηκαν διάφοροι διαδηλωτές οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα από την κοινωνία των πολιτών ε, Αξιβρίσκαν πόδια δηλωτές, με συγχωρείτε. Ε, θα ήθελα να σα παρακαλέσω να το καταδικάσετε δημοσίω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ναι, χθε το βράδυ έγινε μια δημόσια δήλωση από μένα που είχα πει ότι δεν επρόκειτο εγώ να επέμβω να σχολιάζω τι δραστηριότητε των Ευρωβουλευτών. Α περάσουμε τώρα στην επόμενη έκθεση του κυρίου Βό. Δικαιώματα πνευματική διοκτησία στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Έχουμε ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Υπάρχει ένα αίτημα 38 βουλευτών. Τον λόγο έχει η κυρία Ρέγνερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλώ εξ ονόματος των 38 και παραπάνω βουλευτών. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ όλους όσους εργάστηκαν τόσο πολύ για να προστατεύσουν τους καλλιτέχνες και λοιπούς δημιουργούς. Δυστυχώ η οδηγία απαιτεί περαιτέρω ρυθμίσει Την προηγούμενη εβδομάδα το Εθνικό Κόμμα των Εισηγητών ανακοίνωσε δημοσίω πω η οδηγία ω έχει δεν είναι σαφή όσον αφορά τα φίλτρα ανεβάσματο στο διαδίκτυο και είπαν ότι θα τα αποφύγουν αυτά στην εφαρμογή στη Γερμανία. 200.000 άνθρωποι διαδήλωσαν. 5 εκατομμύρια άνθρωποι υπέγραψαν μια αναφορά. Οπότε αγαπητοί συνάδελφοι να υπενθυμίσω ότι ο τίτλος οδηγίας είναι πνευματικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Πρέπει λοιπόν να καθορίζουμε τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες στο ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι στο εθνικό. Γι' αυτό σας παρακαλώ να γίνουν δεκτές οι τροπολογίες και ζητώ να ψηφίσουμε τις τροπολογίες αυτές που έχουν υποβάλει τόσοι πολλοί συνάδελφοι. Σε να παρέμβει ο εισηγητή ή μπορούμε να περάσουμε απευθεία στην ψηφοφορία. Καλώ. Τίθεται λοιπόν σε ψηφοφορία το αίτημα τη κυρία Ρέγνερ με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Επαναλαμβάνω, τίθεται σε ψηφοφορία το αίτημα της κυρίας Ρέγνερ, δηλαδή να ε, γίνουν ε, Γίνουν δεκτές οι τροπολογίες ε, αυτές. Ναι, είναι σαφές το ότι ψηφίζουμε, γιατί υπήρχε μια σύγχυση στις ομάδες. Ψηφίσανε όλοι. Καλώς ε, πέρασε και απορρίπτεται η πρόταση. Ψηφίζουμε τώρα την συμφωνία, την προσωρινή συμφωνία με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Avete votato Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Το κείμενο εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην ε, δήλωση της ε, Κομισιόν. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Με την ίδια νομίζω πλειοψηφία. Λοιπόν, πρώτη ανάγνωση τώρα του Κοινοβουλίου. Ήταν σαφής, είναι η ίδια πλειοψηφία με πριν. Πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου ολοκληρώθηκε. Συγχαρητήρια στον κύριο Φως. νομίζω να τον ε, χειροκροτήσετε ήταν η έκθεση Γκέπχαρτ ε, για το ψηφιακό περιεχόμενο και τις ψηφιακές υπηρεσίες. Περνάμε λοιπόν τώρα στην ονομαστική ψηφοφορία της προσωρινής συμφωνίας. Άρχεται η ε, ψηφοφορία. Πέρας. Το κείμενο εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια και πάλι κύριε Φως και κυρία Γκέπχαρτ. Ψηφίζουμε τώρα την έκθεση αριμών με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Το κείμενο εγκρίνεται. Ολοκληρώθηκε η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Συγχαρητήρια στον κύριο Αριμών. Έκθεση Έγκστρομ Αλληλεία στην περιοχή της Συμφωνίας ΓΙΑΜ. Ψηφίζουμε την πρόταση της Επιτροπής. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Α, με ονομαστική ψηφοφορία. Συγγνώμη. Με συγχωρείτε έρχεται η ψηφοφορία. Έχετε δίκιο. Πέρας. Εγκρίνεται. Δήλωση της ε, Κομισιόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ολοκληρώθηκε η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Συγχαρητήρια στον κύριο Έγκστρομ. Περνάμε στην έκθεση Βάλε ανευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολή εκθέσεων στον τομέα τη περιβαλλοντική πολιτική. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται, ολοκληρώθηκε πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Συγχαρητήρια, κύριε Βαλέαν. Έκθεση Ντέλη. Ειδική κανό για το μέγιστο μήκο των θαλάμων οδήγηση. Προσωρινή συμφωνία. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ολοκληρώθηκε πρώτα ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Συγχαρητήρια κυρία Ντελή. Περνάμε τώρα στην έκθεση Γκίλα. Δείκτες αναφοράς χαμηλών ανθρακούχων. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο. Thank you, Ευχαριστώ. Είχα ε, ζητήσει δύο λεπτά για να μιλήσω, γιατί είναι πολύ σημαντική η ορόσημα η ψηφοφορία. Με βάση τον ΩΣΑ, 6,2 δις ευρώ χρειάζονται παγκοσμίω για να γίνει πιο βιώσιμη η οικονομία μας και να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη στους 2 βαθμούς Κελσίου. Με αυτό κατά νου έχουμε δύο γνώμονες στην έκθεση, ενθαρρύνοντας επενδύσεις να διοχετεύονται ε, σε σχέσεις, ε, σε προγράμματα που περιορίζουν τους ε, τις εκπομπέ άνθρακα για να αποφύγουμε τα προσχήματα υπέρ του περιβάλλοντο και να ευθυγραμμιστούμε με τα κριτήρια των βιώσιμων στόχων ανάπτυξης. Είναι πολυσχεδή βέβαια αυτός ο κλάδος και πολύ συχνά αμελούμε κάποια θέματα. Την πρώτη φορά μάλιστα που έλαβα το λόγο αυτό ήταν όταν ήταν πρόεδρο η κυρία Νικόλ Φοντέν. Έχουν περάσει 20 χρόνια και εξακολουθεί η κυρία Νικόλ Φοντέν να είναι η μοναδική γυναίκα πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάτι μα σοκάρει. Ε, ζητούμε από του παγκόσμιου ηγέτε ισότητα. Πολλέ ε, ε γυναίκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέλαβαν ε, θέση στην Επιτροπή σε Υπουργικά Συμβούλια, αλλά ποτέ δεν είχαμε πρόεδρο ακόμη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είχαμε μόνο μία φορά πρόεδρο γυναίκα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ούτε είχαμε ποτέ γυναίκα πρόεδρο πολιτική ομάδα. Ε, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είμαι στο επόμενο κοινοβούλιο. Θα ήθελα όμω να παρατρύνω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διορθώσει αυτή την ανισότητα και την αδικία. Γιατί από αυτό εξαρτάται η αξιοπιστία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και σίγουρα και στα θέματα της προσέγγισης των περιβάλλοντος μπορεί να ξεπεράσουμε την ανισότητα των φύλων και να κάνουμε το πολιτικό μας σύστημα πιο βιώσιμο και πιο ποικιλόμορφο και πιο πολύμορφο. Ε, δώστε μου λίγο ακόμη δευτερόλεπτα, μπορεί αυτή να είναι η τελευταία μου ολομέλεια. Έχουμε πολλούς ε, παθιασμένου συναδέλφου από πολλούς και το Brexit κατά τη γνώμη μου είναι κολοσιαίο λάθος. Δυστυχώς διακόπτει ο πρόεδρο, Θα ε, πλήξει και τις επερχόμενες γενιέ. Κυρία Γκίλ, ακούσαμε την ε, δήλωσή σας, αλλά πρέπει τώρα να συνεχίσουμε με τις ψηφοφορίε. Κυρία Γκίλ, σας παρακαλώ πολύ. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε δύο προέδρους γυναίκες, την κυρία Κέλλερ και την κυρία Τζίμερ. Είναι παρούσες αυτή τη στιγμή μέσα στην αίθουσα. Προς ενημέρωση σας το λέω αυτό, το ξέρετε δηλαδή. Λοιπόν, ψηφίζουμε την προσωρινή συμφωνία με ονομαστική κλίση. Άρτη η ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρασε. Το κείμενο εγκρίνεται και ολοκληρώνεται έτσι η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Σχαρητήρια, κυρία Γκίλ. Περνάμε στην έκθεση του κυρίου Αριμών. Ειδικέ διατάξει που διέπουν το στόχο Ευρωπαϊκή Δαφική Συνεργασία, Ίντερεγκ. Ο εισηγητή έχει το λόγο. Κύριε Αριμών. Αρημόν, ζητήστε το λόγο, έτσι δεν είναι. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτό το κείμενο και μια ευρεία πλειοψηφία αυτού του ε, Κοινοβουλίου και ομόφωνα η Επιτροπή ζήτησε να στηριχθεί ένα πρόγραμμα μεγάλο όπως το Interreg, ε, το αντίθετο θα λέγαμε του Brexit. Interreg σημαίνει διασυνοριακή συνεργασία με επένδυση ευρωπαϊκών κονδυλίων να κάθονται οι άνθρωποι γύρω από ένα τραπέζι και να βρίσκουν λύσει. Θα ήθελα να λοιπόν ευχαριστήσω του συναδέλφου που εργάστηκαν γι' αυτό και θα ήθελα το Ίντερεγ να λάβει στην επόμενη θητεία τη χρηματοδότηση που το αξίζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ψηφίζουμε αυτή τη στιγμή την ολοκλήρωση εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Αριμόν. Θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων αφρικανικής καταγωγής. Πρόταση ψηφίσματος. Παράγραφος 8, τροπολογία 1, με κλίση άρτη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίσουμε το σύνολο ψηφίσματος με κλίση άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Το κείμενο εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην έκθεση Κόφωτ και Νέντερ Μάιερ. Προβλέπονται πολλές τροπολογίες. Να σηκώντε παρακαλώ πολύ το χέρι κάθε φορά που ψηφίζουμε τροπολογίες. Έκθεση σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή.